Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten anfangen. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε. Ζητώ συγγνώμη από τους ε, καλεσμένους μας για το ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν έρθει τόσοι πολλοί συνάδελφοι. Αλλά ελπίζουμε να υπάρξει μασική προσέλευση ενδιαφερόμενων ακροατών για την απογευματινή μα συνεδρίαση που ελπίζω να είναι πολύ παραγωγική και ελπίζω να ε, μπερδευτεί και κανένα βουλευτής και να μπει στην αίθουσα. Αλλά ας ξεκινήσουμε, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε σήμερα στην ημερήσια διάταξη την ακρόαση για τη νέα τον Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τον Πολιτισμό και έχουμε βεβαίως μια έκθεση ιδίας ε, πρωτοβουλίας από την Κομισιόν τον Απρίλιο, σχεδόν ταυτόχρονα με το πρόγραμμα Creative Europe και βεβαίως αρμόδιος είναι ο κύριος Γραμματικάκης, ο οποίος ελπίζω τουλάχιστον να έρθει. Γνωρίζω ότι είναι κάπου εντός του κτηρίου και ελπίζουμε πραγματικά να συνεισφέρει αυτή η ακρόαση στο να έχουμε μια καλή έκθεση για το ευρωπαϊκό αυτό θεματολόγιο για τον πολιτισμό. Να παρουσιάσω λοιπόν τους προσκεκλημένους μας, να παρουσιάσω τον κύριο Ούγκο Βακέλα, πρόεδρο του Ιδρύματος Φιτς Καράλτο από το Τωρίνο που έχει μια ομιλία με πολύ χαρακτηριστικό τίτλο που ζητάει φιλοδοξία και επαρκή μέσα και το αναμένουμε με αγωνία. Το άλλο έχουμε την κυρία Μέρκελ η οποία είναι επικεφαλής του τμήματος πολιτισμού στην UNESCO της Κολονίας και θα μας μιλήσει για έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο και την επιλογή για πολιτισμικά μέτρα στην Ευρώπη και τέλος η κυρία Ρόζα Πέρες Μονκλού η οποία είναι από εδώ από τις Βρυξέλλες από το Cultural Action Europe και θα μας πει την άποψη της κοινωνίας των πολιτών των ΜΚΟ. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να περιοριστείτε σε 10 λεπτά και μετά από την κάθε παρουσίαση θα έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις και ελπίζουμε να έχουμε ένα παραγωγικό απόγευμα. Θα δώσω τον λόγο πρώτα στον κύριο Βακέλα. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχετε τον λόγο αγαπητέ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Έχουμε ξανασυναντηθεί και έχουμε συζητήσει μεταξύ μας και ελπίζω ότι οι απόψεις μας θα σας δώσουν, θα σας δώσουν κάποιες χρήσιμες ιδέες σφαιρικές. Είχα αποφασίσει να επικεντρωθώ σε μια προσέγγιση μεθοδολογική και κάποιες επιχειρησιακές ιδέες. Επειδή όμως ανησυχώ, όπως φαντάζομαι πολύ και από εσά, ε, λόγω της διάδοσης ε, εκφράσεων και ρητορική που καταλήγουν σε αποτελέσματα, σε ε, υπολοιπόμενα των προσδοκιών μας, συχνά συμβαίνει ε, η πολιτική να ε, παγιδεύονται από τη μια μεταξύ των μεγάλων φιλοδοξιών και των μάντρα που ε, θέλουν να έχουν μια πολύ σφαιρική προσέγγιση που να τα αγκαλιάζει και να τα καλύπτει όλα και χωρίς να ε, σχεδιάζεται δημόσια πολιτική που να βασίζεται σε αποδεκτικά στοιχεία και σε πληροφορίε. Πολλές φορές λοιπόν είναι αντιπαραγωγικό ε, το αποτέλεσμα. Από την άλλη, συχνά ανθεί η βραχυπρόθεσμη λήψη μέτρων κατακαιρματισμένη και χωρίς συγκεκριμένο στόχο, με τομεακές και υποτομεακές ε, προτεραιότητες. Κατά την άποψή μου, αυτές οι πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν το εξής κοινό. Δεν καταλαβαίνουν το βάθος και την πολυπλοκότητα των κοινωνικο-οικονομικών και πολιτιστικών τεχνολογικών αλλαγών. Όλος ιδιαίτερος στη φύση των όσων δρούν και ε, δραστηριοποιούνται στον χώρο της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής καινοτομίας, στην κοινωνία των πολιτών, στα σχετικά κέντρα παραγωγής και στον οικονομικό τομέα. Γιατί λοιπόν οι δημοσίες πολιτικές θα έπρεπε να καταλάβουν πλήρως το φάσμα και σε ό,τι αφορά την, ε, τον πολιτισμό, τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να δημιουργηθούν άειλες και υλικές αξίες πολιτισμός εκπροσωπεί πολύ, διαφορετικ, διαφορετικές δραστηριότητες και τομείς. Και το αφήγημα, ε, έκφραση που χρησιμοποιείται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή για τον τομέα της δημιουργίας και του πολιτισμού, που τους αντιμετωπίζει σαν ένα μεγάλο σύνολο, είναι ένα καλό εργαλείο για να προσπιστούμε τα δικαιώματά τους. οδηγεί σε ωραία δημοσιεύματα στον τύπο, όμως η θάλασσα αυτή της δημιουργίας και του πολιτισμού, γιατί πραγματικά πρόκειται για ένα αρχιπέλαγος, χρειάζεται μια συνολική θεώρηση που να οδηγεί σε δύο επιστημονικές και πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις για την πολιτική και τη χάραξη της και την καινοτομία με συγκεκριμένα στοχευμένα μέτρα πολιτικής, ώστε να ε, καλύπτονται οι αλλαγές, αντί να υπάρχουν παράλληλες τυποποιημένες πολιτικές κονσέρβες. Σήμερα το ενιολογικό πλαίσιο και η εργαλειοθήκη που διαθέτουμε, χάρη στη νέα ψηφιακή οικονομία, συχνά παρουσιάζεται ως η νέα προοπτική για την ανάπτυξη του τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας. Δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα. Ε, διάφορα παραδείγματα από την Ευρωπαϊκή Επικράτεια δείχνουν διαρκώς ότι τα πράγματα ε, προς τα για τον ε, εξής απλό λόγο συντριπτική πλειοψηφία των οργανισμών, των πολιτιστικών ενώ οργανισμών και των οργανισμών δημιουργίας δεν ε, αναπτύσσονται εύκολα με οικονομίες κλίμακας, αγορές κλίμακας και εντατικοποίηση της παραγωγής τους. Ε, τα εκολαπτήρια, οι επιταχύντες, ε, η χρηματοδότηση μπορεί να πηγαίνουν πολύ καλά στον ε, κόσμο των νεοφιών εταιριών τεχνολογίας, αλλά όχι στη δημιουργία και την τέχνη, όπου χρειάζεται χρόνος για να αυξήσει κανείς την παραγωγή του, να αγγίξει μεγαλύτερα κοινά, να παράγει νέες μορφές τέχνης, να αναπτύξει καλλιτεχνικές δραστηριότητες κάποιο, σε κάποια περιοχή. Εάν κοιτάξει κανείς τις πιο ενδιαφέρουσες και νοτόμες δραστηριότητες στον τομέα της τέχνης και της δημιουργίας από τα διάφορα πολιτιστικά ιδρύματα, θα δει ότι πραγματικά αξιοποιούν τις ψηφιακές δημοσιεύσεις αλλά δεν εξαρτώνται ούτε ε, επαφίονται πλήρως την ε, επανάσταση της ψηφιοποίησης. Και δεν είναι ε, σύμπτωση ότι τα οικολαπτήρια δεν λειτουργούν ε, καλά για αυτές τις ε, εταιρείες και τις επιχειρήσεις βιομηχανίας, ε, ναι, συγγνώμη, δημιουργίας, σε αντίθεση με την τεχνολογία. Χρειάζεται οικοδόμηση δυνατοτήτων και όπως κάποιες μελέτες δείχνουν ξεκάθαρα και το τονίζουν, επειδή τα πολιτιστικά ιδρύματα δεν έχουν ε, δεξιότητες management, ούτε την κατάλληλη ε, ομάδα που θα αναλάβει την ηγεσία, δεν μπορούν να αξιοποιήσουν την ψηφιακή επανάσταση για τον πολιτισμό. Πρόσφατα διάβασα μια έκθεση, επικριτική ανάλυση των επενδύσεων, που έχουν πραγματοποιηθεί από κάποια μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα. Έχουν αφιερώσει πολλούς πόρους τον τεχνολογικό του εξοπλισμό. Που όμω ήταν ήδη ξεπερασμένο, Μέσα σε μια διετία ξεπεράστηκε και ήταν παροχημένο. Ε, ε, παροχημένος. Οι λόγοι βάσει της έκθεσης τα αίτια ήταν η έλλειψη δεξιοτήτων, η έλλειψη γνώσης όσων ήταν επικεφαλής αυτών των πολιτιστικών ιδρυμάτων. Γι' αυτό πιστεύω ότι αντί να προστατεύουμε απλώς το περιβάλλον των εταιριών που είναι νεοφύη στον χώρο του πολιτισμού και της δημιουργίας, και εκεί η ατζέντα ε, μπορεί να δώσει κάποιες καλές ιδέες σε προγράμματα. Χρειάζονται διατομεακές πολιτικές που να προωθούν τη συνεργασία και τη συμμαχία μεταξύ των μακροσυμπράξεων επιχειρήσεων με ελεύθερους σκοπευτές ε, στους επαγγελματίες και με ευρύτερης ε, προσέγγισης ιδρύματα, με τη μεταφορά δεξιοτήτων, με τις σχέσεις συνεργασίας. Ε, υπάρχουν κάποια προγράμματα εδώ στην Ευρώπη όπου τα αρχεία, λόγου χαρή, τα μουσεία, χωρίς να κάτσουν να επινοήσουν εξ αρχής τη γνώση, κοιτάζουν πώς να αξιοποιήσουν τις συλλογέ τους και να πολλαπλασιάσουν τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την ψηφιακή επανάσταση. Έχουν αποφασίσει λοιπόν να ανοίξουν τις πόρτες τους με προγράμματα που κρατούν εβδομάδες ή μήνες σε εταιρείε ελεύθερων επαγγελματιών ή μακροεταιρείε για μια νέα γενιά ανθρώπων που θα φέρουν την καινοτομία. Το αποτέλεσμα ήταν ο πολλαπλασιασμός των ευκαιριών, των υπηρεσιών, των ε, ε, προϊόντων και αγαθών και η βελτίωση των υπηρεσιών που παρήχαν αυτά τα πολιτιστικά ιδρύματα. Ταυτόχρονα περισσότερες ευκαιρίες για τις μικρές εταιρείες και όσους έχουν καινοτόμα δράση για να ανταγωνίζονται στη διεθνή αγορά βάσει των προϊόντων που μπορούν να, προτείνουν ε, μέσα από την ευρωπαϊκή κληρονομιά. Οι τρεις τελευταίες μου παρατηρήσεις έχουν να κάνουν με τα πιλωτικά προγράμματα. Νομίζω ότι ιδίω σε καιρού ισχνών αγελάδων θα πρέπει τα ε, προγράμματα αυτά να συμβάλλουν στον δημιουργία ευέλικτων προγραμμάτων και συστημικών αλλαγών, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει μια συνολική διαδικασία αξιολόγησης και διάδοσης των αποτελεσμάτων βάσει μια σειρά αυστηρών προδιαγραφών που να προβλέπονται σε όλα τα επίπεδα. Πρώτη προϋπόθεση. Δεύτερη προϋπόθεση πρέπει να εισάγουμε περισσότερους ποιοτικού δείκτες στην αξιολόγηση. Η ποσοτική καλή είναι, αλλά δεν φτάνουν για να καταλάβουμε και να αναλύσουμε την ποιότητα και την ανάγκη της καινοτομία. Μια άλλη προϋπόθεση είναι να ενισχύσουμε τα ερευνητικά προγράμματα, πράγμα που σημαίνει περισσότερους πόρους, περισσότερα κονδύλια για τα κοινά ερευνητικά κέντρα, διότι πρέπει να έχουμε περισσότερα εμπειρικά στοιχεία, ε, ιδίως για τις διτομιακές περιοχές συνεργασίας. Πρέπει να κατανοήσουμε την αξία και την επίδραση που έχει ο τομέας ε, του πολιτισμού και της δημιουργίας εκτός του χώρου του. Δηλαδή πώς μπορούμε να χτίσουμε γέφυρες ε, μεταξύ του πολιτισμού που θα συμβάλλει στην υγεία, την ευημερία, την κοινωνική συνοχή, δηλαδή σε άλλες περιοχές. Πρέπει να καταλάβουμε τι ε, έχει αποτέλεσμα και τι εταιρείε και επιχειρήσεις θέλουμε να στηρίξουμε. Θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι μια άλλη προϋπόθεση που θεωρώ ουσιώδη και υπ' αυτήν την έννοια μπορεί να κάνει πολλά το Κοινοβούλιο, είναι να στηρίξουμε την διυπηρεσιακή συνεργασία. Έχουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα με το Ευρωπαϊκό Έτος της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπου η συνεργασία μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτισμού και των υπολείπων Γενικών Διευθύνσεων ε, οδήγησε σε άνθεση των δράσεων στους διάφορους, ε, στις διάφορες περιοχές. Αυτό είναι σημαντικό γιατί η διυπηρεσιακή ε, διεπιστημονική αυτή συνεργασία μπορεί να αναπαραχθεί και σε εθνικό επίπεδο πέραν του ευρωπαϊκού και να λειτουργήσει ως καλό παράδειγμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ αγαπητέ για την παρουσίασή σας και τώρα θα δώσω τον λόγο στον εισηγητή μας τον κύριο Γραμματικάκη για τρία λεπτά το πολύ σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η νέα ατζέντα πράγματι αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία ώστε να υιοθετηθεί για πρώτη φορά μια συντονισμένη και ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για τον πολιτισμό. Η πρόταση έρχεται σε μια σημαντική χρονική στιγμή καθώς φέτος διανύουμε το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς το οποίο μας θυμίζει ότι ο πιο σπουδαίος συνεκτικός δρόμος για τους λαούς της Ευρώπης είναι ο πολιτισμός. Αναδεικνύοντας λοιπόν την κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά, ίσως συμβάλλουμε στην πραγματική ενοποίηση της Ευρώπης που σήμερα, το ξέρετε όλοι, υποφέρει από ισχυρές αποσχησιστικές τάσεις. Διαπίστωσα όμως με θλίψη ότι το 36% των Ευρωπαίων, 36% πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν συμμετείχε σε οποιαδήποτε πολιτιστική δραστηριότητα κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Για να αυξηθεί η συμμετοχή, τα κράτη-μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα ώστε οι τέχνε και η δημιουργική σκέψη να συμπεριλαμβάνονται σε όλα τα στάδια τη εκπαίδευση και κατάρτισης. Πρέπει επίση να αυξηθεί και η διασπορά των ευρωπαϊκών έργων τέχνη καθώ και η κινητικότητα των καλλιτεχνών. Η ειδική δράση που προτείνει η Επιτροπή για την κινητικότητα των καλλιτεχνών είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα αρκεί να συνοδεύεται από επαρκή χρηματοδότηση και απλούς στευμένους κανόνες. Θεωρώ επίσης απαραίτητο να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ώστε οι Ευρωπαίοι καλλιτέχνες να μην παραμείνουν βυθισμένοι σε ένα γραφειοκρατικό κικαιώνα. Πρέπει να έχουν απαραίτητη και εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για να εξασφαλίσουν τη στήριξη του έργου τους. Γι' αυτό θα εισηγηθώ στην εισήγησή μου τη δημιουργία μιας ενιαίας φιλικής προς το χρήστη πλατφόρμας που θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με όλα τα διαθέσιμα προγράμματα, αλλά και τις ευκαιρίες επιχορηγήσεων. Θα ήθελα επίσης να χαιρετήσω το γεγονός ότι δίνεται έμφαση στους επιμέρους καλλιτεχνικούς τομείς. Θα σταθώ ιδιαίτερα στην πρωτοβουλία Music Moves Europe, η οποία ευελπιστώ ότι θα ενσωματωθεί, το λέγαμε και παλιότερα, στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη και θα έχει σταθερή χρηματοδότηση. Για την ώρα μόνο το 3% του προγράμματος κατανέμεται στην υποστήριξη της μουσικής και κυρίως βέβαια της κλασικής. Η νέα ατζέντα για τον πολιτισμό παρά τους φιλόδοξους στόχους που θέτει μπορεί να είναι επιτυχής μόνο αν συνοδευτεί από μια σημαντική αύξηση, το υπογραμμίζω, του προϋπολογισμού που διατίθεται στον πολιτισμό, καθώς βέβαια και του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη. Δυστυχώς, παρά τη μεγάλη επιτυχία του, το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη παραμένει υποχρηματοδοτημένο. Αντιπροσωπεύει μόλις το 0,15% του συνολικού προϋπολογισμού και μάλιστα μόνο το 1 τρίτο προορίζεται για τον πολιτισμό. Ενώ η πρόταση της Επιτροπής για την αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη είναι ασφαλώς ένα θετικό βήμα, δεν επαρκεί. Γι' αυτό στην έκθεσή μου σκοπεύω να ζητήσω το διπλασιασμό του προϋπολογισμού μετά το 2020 καθώς και τη δέσμευση των κρατών μελών ότι τουλάχιστον το 1% του επόμενου προπορισμού θα διατεθεί στον πολιτισμό. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σταθώ και στην εξωτερική διάσταση της ατζέντα. Ο πολιτισμός αποτελεί το δυνατότερο όπλο της Ευρώπης. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω σήμερα όλους τους ομιλητές για την συμβολή τους, τη σημαντική, σε αυτή την ακρόαση. Θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω όλα τα σημαντικά σημεία στη συγγραφή της έκθεσής μου, καθώς και στην κατάθεση των σχετικών τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Äh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μια που κάνουμε συνεχώς ε, ερωτοποκρίσεις, θέλετε να πείτε κάτι για αυτό το οποίο είπε ο κύριος Γραμματικά ή όχι. Παρακαλώ. Θέλετε να τοποθετηθείτε ή όχι. Να μείνουμε σε αυτά. Να μείνουμε. Ωραία. Περνάμε στους υπόλοιπους ομιλητές. Η κυρία Τρούπελ. Um, um Σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία η σημερινή ακρόαση για να δούμε το τι θέλουμε πράγματι στο καινούργιο πρόγραμμα. Ήδη συζητήσαμε ότι θέλουμε να υπάρχει μια σαφής ε, διάκριση των προγραμμάτων, δηλαδή ΜΜΕ, πολιτισμός και Music Moves Europe. Να σας δώσω ένα πρόγραμμα. Ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα στο φεστιβάλ του Κάρλο Βιβάρη και μου είπανε, μην το λέτε υποπρόγραμμα ε, media. Δεν είναι, δεν ακούγεται ωραίο τώρα, υπότιτλος και υποπρόγραμμα λοιπά. Χρειάζεται μια καλύτερη στρατηγική επικοινωνίας, θα έλεγα, για να έρθουμε σε επαφή με τους ανθρώπους και ειδικά τους Ευρωπαίους δημιουργούς. Μετά, ναι έχουμε ακριβώς ε, την συζήτηση για τον προϋπολογισμό και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα έχουμε μάχη με το Συμβούλιο, έχουμε ήδη κάποιες ενδείξεις πόσο δύσκολα θα είναι τα πράγματα με τα κράτη-μέλη, αλλά εμεί ω Επιτροπή είμαστε πεπισμένοι κατά ότι πρέπει να δώσουμε αυτήν την μάχη και νομίζω ότι με την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη το θέμα είναι εάν μπορούμε να διατηρήσουμε την έννοια τη ποικιλομορφία στην ε, κοινωνία μας ε, πολιτισμική, θρησκευτική και πρέπει να δούμε ε, και τους διάφορους ανθρώπους. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ε, διαπολιτισμικό διάλογο, συζητήσεις, εκπαίδευση και για εμένα αυτό είναι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα ενωμένη στην πολυμορφία και αν το χάσουμε αυτό και μιλά μόνο για ταυτότητα και ταυτότητες από τα δεξιά και τα αριστερά τότε θα χάσουμε την ψυχή του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Γι' αυτό για μένα είναι τόσο ε, σημαντικό αυτό το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την στήριξή σας. Νομίζω θα συνεργαστούμε τις επόμενες εβδομάδες και πρέπει ακριβώς να έρθουμε σε επαφή με τον ε, κλάδο γιατί πάρα πολλοί κόσμος θέλει να έρθει σε επαφή μαζί μας για το πρόγραμμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και και Βάκελα, θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτό. Όχι, ε, προτιμάω να τα να ακούσω και να κάνω κάποια σχόλια στο τέλο. Μάλιστα. Σίλβια Κώστα για δύο λεπτά. Πραγματικά δεν ήθελα να μιλήσω για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, την οποία είμαι συγγήτρια. Αυτό είναι ένα εργαλείο, ελπίζω, που θα ε, αναλάβει και την ε, ερμηνεία της ευρύτερης ατζέντα για τον πολιτισμό. αυτού του είδους η προσέγγιση με βρίσκει σύμφωνη και χαίρομαι ιδιαίτερος που το είπατε και εσείς προηγουμένως έτσι. Ε, έτσι αναγκαζόμαστε να αναλάβουμε ευθύνε. Διότι δεν πρέπει να χάσουμε τη στόχευση και να εξοπλιστούμε σωστά. Διότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια ατζέντα για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό ε, με βάση τα όσα πρόκειψαν από την τελευταία δεκαετία και ίσω για τα επόμενα δέκα χρόνια, για το μέλλον πάντω, και να είμαστε συνεπεί και με του στόχου τη ατζέντα και τα εργαλεία που ε, θα προβλέπει και με τι πολιτικέ, μια πώληση για την ευρωπαϊκή κουλτούρα που θα προβλέψουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ε, επειδή ε, δεν θα πρέπει τα εργαλεία της Δημιουργική Ευρώπης, του Creative Europe, να είναι λιγότερο στοχευμένα από αυτά που προβλέπουμε στην ατζέντα αυτή. Ε, τώρα, αυτά που θέλω να πω. θα θέλαμε λίγες περισσότερες λεπτομέρειες, για το ότι δεν θα πρέπει να μαγευτούμε από μια λύση ψηφιακή που θα μας αγινεύσει τελείως και θα ξεχάσουμε τα υπόλοιπα. Πρέπει να έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία και για τις ψηφιακές επιχειρήσεις, ναι, αλλά δεν θα είναι αυτή η μόνη κατάλληλη λύση για τι μικρέ, μικρότατε επιχειρήσει και όχι μόνο επιχειρήσει, αλλά πολλέ φορέ ενώσει και με κυβερνητικέ οργανώσει, οι οποίε θέλουν να αναπτυχθούν. Θέλουν να αναπτυχθούν και να αναπτύξουν προϊόντα και καινοτόμε υπηρεσίε, αλλά και προϊόντα για την πολιτιστική κληρονομιά. Ε, αυτό είναι σημαντικό. Σε σχέση με αυτό το σημείο, λοιπόν, και επειδή θα είδατε το πρόγραμμα τη Δημιουργική Ευρώπη και ε, ελπίζω με σχέση, σε σχέση με την πολιτική που έχουμε εφαρμόσει τα τελευταία χρόνια με την ε, πολιτιστική διπλωματία διεθνώ, με την πολιτική για τι μικρέ και μικρότατε επιχειρήσει στον χώρο τη δημιουργία και της, ε, του πολιτισμού, με τη στρατηγική για τι δεξιότητε. Θεωρείτε ότι έπρεπε να δώσουμε διαφορετικό προσανατολισμό στι προτεραιότητέ μα. Νομίζω από την ομιλία σα προέκυψε ότι πρέπει να επενδύσουμε στα πρόσωπα, στου ανθρώπου. Σε αυτού που είναι καινοτόμοι οι ίδιοι και όχι απλώ στη λέξη και τον όρο καινοτομία έτσι θεωρητικά και αφηρημένα. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να πω. Και θα ήταν ενδιαφέρον να ε, ε, ξερευνήσουμε και τους τρόπους. Θα μπορούσαμε ίσως να δημιουργήσουμε hub δεξιοτήτων, ε, κομβικά σημεία δεξιοτήτων, όχι μόνο για τα κολαπτήρια νέων εταιριών και δραστηριοτήτων. Ναι, να μιλήσω ταλικά. Νομίζω ότι κέντρο του ενδιαφέροντό μα θα πρέπει να είναι όντω οι άνθρωποι, τα πρόσωπα. Θα πρέπει να καταφέρουμε να φέρουμε πραγματική καινοτομία, όχι ένα νέο πρόγραμμα, όχι ένα νέο είδος εφαρμογής με διαφορετικά μέσα, αλλά την πραγματική τεχνολογική ψηφιακή εθνική επανάσταση να τη φέρουμε στο κέντρο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Δεν μπορεί το μέλλον της παραγωγής, διανομής και πρόσβασης στα πολιτιστικά να ε, ανατίθεται απλώς με όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται έστω και με εξαιρετικό τρόπο ως τώρα, να προέρχονται από την παραδοσιακή ιστορική ε, υποδομή και εγκατάσταση των πολιτιστικών ιδρυμάτων. Διότι έχουμε κάποια ιδρύματα που έχουν πάρει μια προδιαγεγραμμένη πορεία με, περισσότερο, με περισσότερες ή λιγότερες δυνατότητες να αντιληφθούν και να προσελκύσουν την καινοτομία και η πραγματική παραγωγή προκύπτει εκτός των ιδρυμάτων αυτού, εκτός του πεδίου δράσης τους. Υπάρχει και κίνδυνος ως προς την, τις γενιές, το γενελογικό χάσμα. Εάν δεν καλλιεργήσουμε τη δημιουργία προϋποθέσεων για να πάμε στην παγκόσμια αγορά, η ευρωπαϊκή αγορά, που ε, εξασφαλίζει συνθήκες στην αγορά με βιωσιμότητα ε, και ε, κερδοφορία στις μικρότατες, μικρές επιχειρήσεις που θέλουν να λειτουργήσουν και να πτήσουν σε αυτό το πεδίο, θα βγουν από το χώρο του πολιτισμού, διότι αν δεν έχουν καμία προοπτική στην αγορά, μια καινούργια, μια νεοφύση εταιρεία, το λέω, επειδή έχω εργαστεί ε, στο διοικητικό ε, τέτοιων μικρών επιχειρήσεων, πάνε σε άλλο χώρο, στα χημικά, στα φάρμακα. Εκεί βρίσκουν κονδύλια, βρίσκουν επενδύσεις. Μισό εκατομμύριο ευρώ, γιατί μπορεί να φέρουν ένα κέρδος 5 εκατομμυρίων στον επενδυτή. Ε, διότι δεν φαντάζεται κανείς ότι ξέρω εγώ, η βελτίωση πρόσβασης σε ένα μουσείο θα δεκαπλασιάσει την αρχική του επένδυση ο επενδυτής δεν θα έχει την ίδια κερδοφορία μέσα σε μια τριετία από ότι, σε σύγκριση με ό,τι μπορεί να συμβαίνει στον χώρο της τεχνολογίας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα περνάμε στον δεύτερο, στην δεύτερη προσκεκλημένη μας, την κυρία Μάρκελ, όπως σας είπα, επικεφαλής του Τμήματος Πολιτισμού και Σκέψης για τον Κόσμο στην UNESCO της Κολονίας και χαίρομαι που θα σας ακούσουμε. Έχετε τον λόγο. Για δέκα λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσω και εγώ στα αγγλικά. Εξετάσαμε πολύ προσεκτικά και την ανακοίνωση της ε, Κομισιόν και το έγγραφο εργασίας που περιέχει πολλά εμπειρικά στοιχεία και είναι πράγματι ένα ε, ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει μια δυναμική για να έχουμε ένα συνολικό πλαίσιο για τα μέσα και τις πλατφόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πράγματι όπως λέει το άρθρο 167 το θέμα είναι ακριβώς ο σεβασμός του πολιτισμού και η ποικιλομορφία και ακριβώς το θέμα του χρονικού ορίζοντα είναι κάτι ενδιαφέρον. Είναι το 2030, είναι το 2050. Οπότε βλέπουμε και την δική μας εμπειρία από τη Γερμανική Επιτροπή της UNESCO και την Διεθνή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως εστιάζουμε στο τι είδους δημοσία πολιτική απαιτείται σήμερα στον τομέα αυτών. Γι' αυτό έχω εστιάσει σε τέσσερα στοιχεία. πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι ε, επιλέχθηκε να ξεκινήσουμε με την πολιτιστική συμμετοχή και την αντίληψη το ποιος είναι ο ρόλος του πολιτισμού αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Δεύτερον, εκτιμούμε το ότι έχουμε φέτος το ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς. Τρίτον, κοιτάω λίγο το στοιχείο της κινητικότητας που έρχεται έτσι πολύ δυναμικά. Και τέλος, η έννοια του ευρωπαϊκού πολιτισμικού χώρου και οι σχετικές ε, λεπτομέρειες. Να ξεκινήσω λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον είδαμε τα δεδομένα του Ευρωβαρόμετρου και κάποια άλλα δεδομένα που αναφέρατε ήδη εσείς, η συμμετοχή δηλαδή σε πολιτισμικές δραστηριότητες, είναι ένα ε, πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Δηλαδή κοιτάμε το 66% που συμμετέχει ή τους μη συμμετέχοντες και εκεί πέρα ακριβώς έχουμε και τα στοιχεία της πιο πρόσφατης έκθεσης της UNESCO του 2016 και εκεί πέρα θα προσπαθήσω να διευρύνω λίγο το φάσμα να δω πού βρισκόμαστε. Γιατί οι δείκτες αυτοί είναι εντυπωσιακοί, αλλά εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να σκεφτούμε και τρεις διαστάσεις ακόμα υπάρχουν πολλές ε, αυτοοργανωμένες, όπως λέγονται, πολιτισμικές πρακτικές, ε, ζωντανή κληρονομιά, αλλά και σύγχρονη έκφραση. Παραδείγματος χάρη στην χώρα μας έχουμε 20 εκατομμύρια μέλη σε διάφορες ενώσεις ε, που αυτοοργανώνονται και βλέπουμε αυτό το οποίο είχαμε τον κλασικό πολιτισμικό χώρο που εξελίσσεται. Οι χώροι εξελίσσονται σε υβριδικούς χώρους και συνδέουν τα ΜΜΕ με τους πόρους. Παράδειγμα τους κάνει οι δημόσιες βιβλιοθήκες. 100 εκατομμύρια άνθρωποι πηγαίνουν σε αυτές τις βιβλιοθήκες ε, ε, κάθε χρόνο. Είναι ο ίδιος αριθμός ε, των ανθρώπων που πάνε στο γήπεδο. Και ακριβώ αυτό το είδαμε στην παγκόσμια έκθεση της UNESCO να ρωτήσουν τον κόσμο ποια είναι η σημαντική τους ε, πολιτισμική δραστηριότητα και το βασικότερο να τον κόσμο είναι να βλέπουν τηλεόραση και να ακούν ραδιόφωνα και για τα παιδιά γνωρίζουμε είναι το βίντεο. Είναι μια πολύ σημαντική έκθεση. Οπότε έχουμε κάποια διασυνδεδεμένα λοιπόν οικοσυστήματα. Οπότε έχουμε ένα πρώτο συμπέρασμα. Έχουμε λοιπόν ένα πλαίσιο το οποίο αλλάζει αυτή την στιγμή και η καινοτομία στον πολιτισμό είναι ε, ένας χρήσιμος όρος, οπότε θα θέλαμε το Κοινοβουλίο να επεκταθεί επ' αυτού και πράγματι η δίκαιη αμοιβή των καλλιτεχνών και των δημιουργών σε αυτό το πλαίσιο ε, παίζει ένα ρόλο κλειδί, αν θέλετε, να έχουμε το ίδιο τοπίο σε 10 χρόνια από σήμερα. Η δεύτερη σύσταση είναι πράγματι να επανεξετάσουμε ακριβώς αυτή την έννοια της συμμετοχής στον πολιτισμό και να μην συνδέουμε μόνο αυτά τα τρία οικοσυστήματα που ανέφερα αλλά και την σχέση μεταξύ της ποικιλομορφίας των ΜΜΕ και της πολιτισμικής έκφρασης. Δεύτερο και θα επιταχύνω λίγο, ήδη ακούστηκαν αρκετά για το πόσο δυναμική είναι η ιδέα του πολιτιστικής κληρονομιάς. Ε, είχαμε παραδείγματο χάρη μία εστίαση στην δομημένη παρουσίαση και υπήρχαν βεβαίως και οι αντιδράσεις από ανθρώπους, από βιβλιοθήκες, συντρίμματα κτλ. Και η Γενική μας Συνέλευση επίσης πρόσφατα το ξαναείδε αυτό και είπαμε ότι θα πρέπει να είμαστε κάπως πιο φιλόδοξοι, δηλαδή τι εννοούμε και τι κρύβεται πίσω από τα μνημεία επίσης, γιατί συχνά υπάρχει ακριβώς η το θέμα του πολιτισμού, της δημιουργίας του πολιτισμού που περιέχει αρκετά μεγάλη κινητικότητα η οποία δεν φαίνεται και ακριβώς έτσι προχωράμε και με το ευρωπαϊκό οικοδόμα αλλά και σύνδεση με άλλα μέρη του κόσμου γιατί πολλές από αυτές τις ταυτότητες είναι πολλαπλές, υβριδικές και ε, αλλάζουν σε όλη την ιστορία και θα συνεχίσουν να αλλάζουν. Αναφέρθηκε ο Αμάρτια Σεν και καλό θα ήταν να το εμβαθύνουμε νομίζω αυτό. Και Κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ των όσων κάνουμε στο εσωτερικό και των όσων σκεφτόμαστε ως ο πολιτισμός της διεθνής σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί βεβαίω ε, αυτά τα δύο συνδέονται. Δύο στοιχεία ακόμα. Ναι, η κινητικότητα έχει ε, σημασία, είναι ένα στατικό προαπαιτούμενο για να προωθήσουμε την συνδημιουργία και όλα τα στοιχεία αυτά στο σχέδιο είναι πάρα πολύ σημαντικά και αφορούν και την πρακτική εφαρμογή, το πώς δηλαδή θα υπάρχει μια διυπουργική συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με το Υπουργείο Εσωτερικών ή κάτι άλλο. Και ακριβώς ε, εδώ πέρα θέλουμε υλοποιήσιμες προτάσεις. Η πιλωτική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Κινητικότητας είναι πολύ χρήσιμη και σας παρακαλώ να θυμάστε ότι ε, το ζήτημα αυτό δεν είναι μεμονωμένο, είναι στο πλαίσιο μιας ευρύτερης δέσμευσης όλων των κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως περιφερειακού οργανισμού, γιατί βεβαίως αυτά τα είχε πει ε, ακριβώ και η σύμβαση της UNESCO που στόχο έχει να διευκολύνει ακριβώς την ροή και την κινητικότητα των καλλιτεχνών ως ένα είδος προτιμησιακής μεταχείρισης θα έλεγα και νομίζω ότι καλό θα ήταν να αναπτύξουμε νέες ιδέες ως προς αυτό. Είναι πολύ ενθαρρυντικό αλλά χρειάζεται και κάποια διευκρίνηση το αν μπορεί να χρηματοδοτηθεί αυτό από το Erasmus Plus, Erasmus ε, Culture, ε, πώς, όπως και να το πούμε, αλλά είναι μια επένδυση σε βάθος χρόνου. Τέλος, η έννοια του ευρωπαϊκού πολιτιστικού χώρου είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για να επανενωθεί η Ευρώπη εκ των έσω. Και ακριβώς έχουμε μάθηση μεταξύ ομοτήμων, μεταξύ κοινοτήτων, χρηστών και έχουμε και ενδιαφέρουσες εμπειρίες στο επίπεδο της πόλης. Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα να υπάρξει μια κινητοποίηση για να ξεπεράσουμε ακριβώς κάποιες από τις λανθασμένες ε, διαχωριστικές γραμμές που βλέπουμε και όπως είπε και ο κύριος γραμματικά ναι πράγματι και οι λεπτομέρειες οι πρακτικές έχουν σημασία και όσο πιο δυσκίνητα είναι τα πράγματα τόσο μεγαλύτερη θα είναι η συνεργασία ή να μην αντιμετωπίζουν γραφειοκρατικά εμπόδια οι δημιουργεί. Οπότε το θέμα είναι ακριβώς να οθηθεί η δυνατότητα μάθησης της νέας γενιάς των ανθρώπων που δημιουργούν στην Ευρώπη. Αυτή είναι, αν θέλετε, η ευκαιρία και το διακύβευμα. Οπότε, ναι, η πρόταση για μια νέα ευρωπαϊκή ατζέντα πολιτισμού είναι επίκαιρη, είναι μια επίκαιρη πρωτοβουλία για τα οικοσυστήματα αυτά της πολιτισμικής πολιτικής και καλό θα είναι ακριβώς να συνδέσουμε τα σχετικά αυτά στοιχεία και να ενθαρρύνουμε την εσωτερική και την εξωτερική διάσταση. Γιατί υπάρχουν βεβαίως και πολλές προσδοκίες από την Ευρώπη σε ολόκληρο τον κόσμο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και βεβαίως η ε, σε αυτό θα γίνει μέσω της UNESCO και άλλων οργανισμών γιατί βρισκόμαστε σε μια φάση μετασχηματισμού και δεν το γνωρίζουμε αλλά ελπίζουμε να καταλήξουμε με τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό μιας βιώσιμης ανάπτυξης στο ψηφιακό πλαίσιο που είναι το δημοκρατικό καθήκον και πρόκληση του καιρού μας. Ε, Σα ευχαριστώ λοιπόν και αναμένω τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και για την εκτίμηση την οποία κάνατε. Δεν βλέπω κάποιον να ζητάει τον λόγο. Θα μιλήσω λοιπόν εγώ. Στη Γερμανία το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο που εκπροσωπούνται τα κρατήδια ε, είχε μια γνωμοδότηση η οποία δεν ήταν και πολύ αισιόδοξη θα αναφέρω ένα σημείο που θεωρώ ότι πραγματικά ε, είναι επίκαιρο και πείτε μου αν συμφωνείτε. Λένε εκεί πέρα ότι λυπούνται για την κατεύθυνση της πολιτικής ε, πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που εξακολουθεί να είναι υποτεταγμένη σε μία αντίληψη χρήσιμοθυρική ενώ θα έπρεπε να έχει ως στόχο μία πλούσια και ποιοτική προσφορά πολιτισμού και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη του πολιτισμού, κάτι το οποίο δεν φαίνεται καθόλου στην πρόταση της Κομισιόν και συνεχίζει ότι ο προσανατολισμός στους τρεις στρατηγικούς στόχους ε, ε, είναι κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερο συστατικό και μάλιστα λέει ότι η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου αντικαθίσταται από την κοινωνική διάσταση του πολιτισμού και περνάει σε δευτερεύοντα ρόλο η πολιτισμική ποικιλομορφία και ο διαπολιτισμικός διάλογος και απορρίπτουν αυτήν την ιδέα του πολιτισμού ως πόρου, εάν θέλετε. Εντάξει, ε, βεβαίως οι χώρε ε, λένε μεν ότι μακριά τα χέρια από τον ε, πολιτισμό είναι δική μας αρμοδιότητα, αλλά βλέπουμε ότι η Γερμανία λέει ότι θα έπρεπε να πάει προς μια άλλη κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ερώτηση, γιατί διάβασα αυτό με μεγάλη προσοχή θεωρώ ότι ε, έχει κάποιο δίκαιο εδώ πέρα το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Γερμανίας γιατί ε, είναι ξεκάθαρο και στο έγγραφο της Κομισιόν από την διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους 82% λένε ότι χρειαζόμαστε αυτόν τον στόχο υπάρχει στην ε, συνθήκη αλλά εάν δεν το λέμε καθαρά την πολιτισμική πυκλομορφία και του διαλόγου για τις διαφορές ε, αυτό είναι το, το βασικό. Και από αυτήν την έννοια ε, θα ήθελα να ζητήσω ακριβώ να το ξαναδείτε αυτό από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Μια εγκάρσια διάσταση ή ως ε, στόχος το πώς θα διατυπωθεί είναι ένα ερώτημα, αλλά ίσως να είναι θέμα και παρεξήγηση το τι εννοούμε εδώ πέρα δηλαδή χρήσιμο και χρησιμοφυρία. Δεν διάβασα την ανακοίνωση. Είδα αυτό ακριβώς ότι θα έπρεπε να περιέχεται πολύ περισσότερο αυτή η διάσταση της κινητοποίησης των πολιτών σε σχέση με πριν από 10 χρόνια, γιατί έχουμε μια νέα κατάσταση με μεγάλες προκλήσεις στην Ευρώπη, αλλά Θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτήν την ε, ερώτηση γιατί θα έλεγα ότι μπορεί πράγματι να είναι ενδιαφέρον ότι ε, πρέπει να το δείτε αυτό στο πλαίσιο της έκθεσης σας. Δηλαδή είναι ένα θέμα είτε το ένα είτε το άλλο. Γιατί ε, λέμε και στα αγγλικά η πολιτισμική πόρη ε, δεν σημαίνει μια ε, χρησιμοθυρική αντίληψη σημαίνει οτιδήποτε. Το ότι μπορεί να διδάσκεται με κάποια συγκεκριμένα τεχνικά μέσα, η τέχνη κτλ. Και ακριβώς θεωρώ ότι η εστίαση στην κινητικότητα είναι ακριβώς κατάλληλη αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα και διαφορετικά, έτσι ώστε οι επαγγελματίες, ή καλλιτέχνες, αλλά και παραδείγματος χάρη και οι αρμόδιοι σε πόλεις, σε περιφέρειες, να συνεργαστούν πέρα από τις ε, συναντήσεις της Βρυξέλλες και θεωρώ ότι είναι μια σωστή κατεύθυνση που θα πρέπει να ενισχύσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χέλγα Τρίπελ Ναι, ενδιαφέρον αυτό το οποίο είπε η κυρία Μέρκελ. Δηλαδή έχουμε την κινητικότητα και ακριβώς ε, την επαφή έχουμε αυτή την πολιτική συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου αποφασιστικό είναι ακριβώς το εάν θα καταφέρουν οι φιλελεύθερες δημοκρατίες να το ξεκαθαρίσουν αυτό το πράγμα. Βεβαίω ε, τίθεται και το ζήτημα ακριβώς ε, του αν ε, το διαφορετικό θα επιβληθεί ή θα το επιβληθούμε. Βεβαίω εντάξει, ζω σε μια κοινωνία που όλοι είναι ε, διαφορετική από εμένα. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι αυτό το πνεύμα, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και αλλού, ε, υπονομεύεται και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε να γίνει αυτό. Ζούμε από την πολιτισμική ε, ποικιλομορφία. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό να το τονίσουμε αυτό, ότι το θέλουμε αυτό το πράγμα. Τώρα εγώ αυτό το ερμηνεύω αν θέλετε, γιατί εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να καλυτερεύσουμε το κείμενο της Κομισιόν, αλλά θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα, γιατί ανησυχώ. Πριν από δύο χρόνια είχα βγάλει ένα, μια ομιλία και εκεί πέρα ακούστηκε ακριβώς το ότι ε, πρώτα απ' όλα υπάρχει στην αρχή αυτής της αλυσίδας δημιουργίας της πολιτισμικής αξίας υπάρχει το δημιουργικό σκέλες ε, και βεβαίω ε, πρέπει να δούμε και το ότι οι νέοι πράγματι ενδιαφέρονται για τις θέσεις εργασίας, χημικές βιομηχανίες, τα αυτοκίνητα. Αλλά δεν είναι κάτι το ξένο ή δημιουργικές, ε, ο δημιουργικός κλάδος. Και βέβαια η κυρία Μέρκελ το είπε, δεν είναι μόνο τα λάθος κριτήρια της χρησιμοθυρίας και να λέμε όχι, ναι, αυτά είναι νεοφιλελεύθερα, οικονομία στον πολιτισμό κτλ. Όχι, εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο στην τελευταία έκθεση της Κομισιόν, αλλά ο πολιτισμός ως πόρος, εάν δούμε ακριβώς το θετικό, τη θετική του πτυχή και όχι ως κάτι το περιθωριακό, είναι ακριβώς κάτι το οποίο λέμε ότι είναι σημαντικό. Διάλογος, ε, διαφορές ε, και τα λοιπά. Αυτό το αντιλαμβάνομαι εγώ, αυτό το οποίο λέμε ως πόρος ε, στα αγγλικά. Ε, έτσι, το θεωρώ κάτι το καλό, κάτι το θετικό. Εκτός εάν βεβαίως κάποιοι χρησιμοποιούν τον πολιτισμό μόνο για να υπάρξει μια αντιδημοκρατική περιχαράκωση. Υπάρχει βεβαίως και αυτή η κατάχρηση. Γνωρίζουμε αυτή την εθνικιστική τάση ε, βλέπουμε κάποια παραδείγματα εντό και εκτός της Ευρωπαϊκή Ένωσης, αλλά ε, εμείς πρέπει να τα αφήσουμε προς μια δημοκρατική πολιτισμική αντίληψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Μέρκελ, θέλετε να πείτε κάτι. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο είδαμε στο ευρωβαρόμετρο που είχα μια ξεκάθαρη ε, στήριξη του ευρωπαϊκού εγχειρήματο στο κομμάτι που έλεγε τι είναι αυτό το οποίο συνδέει τους Ευρωπαίους πολίτες και τα βασικά ήταν ε, πολιτισμός, ιστορία και αξίες. Αυτό το πρόγραμμα επίσης, το Memory of the World της UNESCO όπου συνεργαζόμαστε οι Ευρωπαίοι και είναι μια διάσταση που ήθελα να τονίσω ότι έχουμε μια αρκετά ευρύτερη κοινότητα που υπάρχει οπότε έτσι ακριβώς έχουμε αυτές, αυτά τα, τα, τις τρεις βασικές ελευθερίες ε, την καλλιτεχνική, την μηντιακή και την επιστημονική ελευθερία και έτσι νομίζω αυτά κάνουν τις κοινωνίες ε, παραγωγικές ε, και δυναμικές. Οπότε έχουμε αυτό το οποίο είπε το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο. Ε, θα πρέπει να το δούμε υπό αυτό το πρίσμα και στην έκθεσή σας νομίζω ως Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σιλβία Κώστα. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο διάλογος. Μας βοηθάει να καταλάβουμε. Παρακαλώ τα ακουστικά σας. Είναι σημαντικός αυτός ο διάλογος μεταξύ μας. Καταλαβαίνουμε πού πρέπει να στοχεύσουμε, σε ποιε πτυχέ που φαίνεται ότι δεν φωτίζονται συνήθω αρκετά. Χρήσιμη ανταλλαγή. Επ' αυτού, να πω ότι μπορεί, μπορεί οι τρει στόχοι που έχουν ονομαστεί κοινωνικοί δεν αφήνουν να αναδειχθεί αυτό που είναι σημαντικό. Τρεις λέξεις. Κοινή πόρη, αξίες που ενισχύουν και η ε, κοινή ιστορία. Αυτά εξηγούν ε, την ουσία του προγράμματος ε, για την Ευρώπη. Η ελευθερία όμως της καλλιτεχνικής έκφρασης και της δημιουργικότητας των ανθρώπων, των δημιουργών, ως πόρος πολιτιστικής καινοτομία είναι κάτι σημαντικό. Ίσως θα πρέπει να γίνει πιο σαφές. Και ήταν ενδιαφέρον αυτό που είπατε εσείς για τη σχέση συνέπειας μεταξύ των εσωτερικών δράσεων και των εξωτερικών Ίσως να το αναλύαμε κάπως καλύτερα, διότι παρακολούθησα και την υλοποίηση της στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Διπλωματία. Υπάρχει και ένα τρίτο σκέλος εδώ. Είναι σωστό τα στοιχεία αυτά του διαπολιτιστικού διαλόγου και του, πώς να το πω, του πώς εξάγουμε την Ευρωπαϊκή τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, αλλά όχι μόνο, όπως μπορούμε να είμαστε ευρωπαϊ... Ε, πολιτιστικοί πρωταγωνιστές στον κόσμο. Και αυτή είναι μια σημαντική νέα πρόκληση. Ενδιαφέρει ακόμα και την UNESCO, ε, UNESCO συγγνώμη, και θα πρέπει και εσείς να έχετε από αυτού κάποια άποψη. Ευχαριστούμε Σιλβία. Κυρία Μέρκελ. Θα απαντήσω στα αγγλικά. Το ζήτημα είναι ότι το άνοιγμα των εθνικών αγορών και των δυνατήτων παραγωγής όντως είναι προς το συμφέρον μας, πράγματι γιατί εμπλουτίζει την προσφορά των χωρών μας και γίνεται μια πραγματικότητα έτσι κι αλλιώς. Πριν από 10 χρόνια οι στόχοι μπήκαν σε ένα πλαίσιο παγκοσμιοποίησης. Δεν ήταν όπως σήμερα. Αν δούμε πώς λειτουργεί ο χώρος του πολιτισμού και της τέχνης, βλέπουμε ότι από τις επαγγελματικέ κοινότητες μέσα αρχίζουν να αναπτύσσονται διάφορες λύσεις. Έχουμε δουλέψει μεταξύ των μεσογειακών χωρών, για παράδειγμα, υπάρχει ανταλλαγή στην Μεσόγειο. Ο τρόπος που γίνονται τα πράγματα σήμερα είναι αλλιώ και είναι πολύ καλύτερα αν μαζί τα κάνουμε και τα βάζουμε σε ένα πλαίσιο αντί να τα χωρίζουμε σε τομεί, σε κλάδου. Η κινητικότητα λοιπόν και η πολιτική φιλοδοξία που έχουν όλες οι χώρες μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να πουν όλα στο ίδιο επίπεδο και πιστεύω ότι είναι εφικτό θέλουμε περισσότερη δικαιοσύνη στην έννοια του πολιτισμού. Όταν μιλάμε για ελεύθερη αγορά, είναι κάτι εφικτό. Στη μουσική, για παράδειγμα, υπάρχει μεγάλος δυναμισμός. Οπότε αναγνωρίζω πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία και στους στόχους και στο έγγραφο που δείχνουν ότι μεταξύ ομολόγων σε επαγγελματικό επίπεδο τα πράγματα έχουν εξελιχθεί πολύ. Θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες και στην έκθεση της UNESCO. Η κινητικότητα έχει ενισχυθεί. Οι Ευρωπαίοι επαγγελματίες βέβαια έχουν διπλές δυνατότητες από αυτές που έχουν ε, οι δημιουργοί στα άλλα μέρη του κόσμου. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε στο επόμενο. για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Βόρτ. Πολύ θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η γνώμη του πάνελ για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης που δεν είναι στους ε, πολιτιστικούς στόχους. Όταν μιλάμε για τις ευρωπαϊκές αξίες και για τη δημοκρατία, όταν μιλάμε για την ε, σημασία που έχει να καταλάβουμε ο ένας τον πολιτισμό και την οτροπία του άλλου και ότι θα μας βοηθούσε αυτό να καταλάβουμε που βρισκόμαστε, ε, θα έπρεπε ρητά να το λέμε ότι είμαστε υπέρ της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και εμένα με απασχολεί πολύ το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνεται στους στόχους. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Merkel. Καταλαβαίνω και εγώ ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρουμε ήδη τις λεπτομέρειες. Αν το συγκρίνουμε με τις συνολικότερες εκθέσεις για την αναδιαμόρφωση της πολιτικής και δούμε τις θεμελιώδεις ελευθερίες, η ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης ε, και η ε, ελευθερία που, και οι ελευθερίες που αφορούν ε, τα, την ταυτότητα του φίλου είναι οι βασικές είναι οι τρεις βασικές ελευθερίες που συνδυάζονται καλλιτεχνική, επιστημονική και προσωπική. Και οι τρεις ε, ε, αλληλεπηρεάζονται και επιτρέπουν στον τομέα των μέσων, είτε ανήκουν στο δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε στο διαδίκτυο, να ε, προχωρήσουν. ένας γάμος που γίνεται κάπως φυσικό το τρόπο, για να το πω έτσι. Είναι ένα τέταρτο οικοσύστημα που αναπτύσσεται. Έτσι πρέπει να το σκεφτόμαστε, ειδικά αν το σκεφτόμαστε όπως είπατε. Αυτά. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω κι εγώ. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα την άποψη της ε, κοινωνίας των πολιτών και την κυρία Ρόζα Περές Μονκλού από το Cultural Action Europe. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας να συμμετάσχω και εγώ σε αυτή τη σημαντική ακρόαση εκ μέρους της Culture Culture Action Europe. Εμείς δουλεύουμε για το μέλλον των ευρωπαϊκών πολιτικών. Εδώ και 1,5 χρόνο είχα μια παρουσίαση, δεν ξέρω αν τη βλέπετε. Λοιπόν, η εντολή μας ποια είναι. Είναι ο πολιτισμός να μπει στην καρδιά της εκπόνησης πολιτικών. Και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι δουλεύουμε με τα μέλη μας, με τους εταίρους μας, με τους πολίτες, με όσους εκπονούν πολιτική, για να ακούμε και ποια είναι η δικιά τους η γνώμη όσον αφορά το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολιτικής. Σήμερα θα σας παρουσιάσω μια αξιολόγηση λοιπόν για το πώς εκτιμώνται οι σημερινοί στόχοι. Να σας πω πρώτα τι είναι η Culture Action Europe. Είναι ένα δίκτυο δικτύων, είναι μια κοινότητα που αποτελείται από διεθνή και εθνικά δίκτυα από όλους τους πολιτιστικούς κλάδους, είτε πρόκειται για τη μουσική, για το χορό ε, και ε, συμμετέχουν επίσης και πολιτιστικές οργανώσεις, ιδρύματα και άτομα μεμονωμένα. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε ποια είναι τα διάφορα ζητήματα και ποιες είναι οι τάσεις και να δούμε στη συνέχεια τι γίνεται στο μέλλον. Είμαστε λοιπόν μια κοινότητα. Συμμετέχουμε στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό χώρο. Μερικές φορές είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Μοιάζει σαν αυτό που βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια. Εδώ βλέπουμε τις διασυνδέσεις μεταξύ των μελών της οργάνωσής μας, της Culture Action Europe και των μελών. Δεν είναι πάντα εύκολο να μετρήσει κανείς και να υπολογίσει ποιες είναι οι επιπτώσεις της πολιτιστικής πολιτικής. Παρόλο που η εικόνα πολλές φορές είναι πιο ισχυρή από τις λέξεις, από τα λόγια. Είμαστε λοιπόν ένα πολύ όμορφο οικοσύστημα διασυνδέσεων. Και τι συμβαίνει μέσα σε αυτή την κοινότητα, κυκλοφορούν ιδέες, δημιουργούνται συνεργασίες, εταιρικές σχέσεις και επίσης κοινή δράση. Σήμερα πρέπει να υπογραμμίσω ότι όλα αυτά είναι χάρη στην πολιτιστική πολιτική, που έχει βέβαια αυτή την ε, περίπλοκη μορφή και γιατί, γιατί το ευρωπαϊκό μοντέλο αποφάσισε να δώσει μεγάλη σημασία στην πολυμορφία. Αποφασίσαμε να συζητάμε με όλους. Αλλιώς θα είχαμε κάτι πολύ πιο απλό εδώ, θα ήταν πιο απλή αυτή η εικόνα. Γι' αυτό λοιπόν οι στόχοι για τον πολιτισμό και σημερινή συζήτηση έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπημένη πολιτική και την είχαμε μέχρι τώρα και αυτό βοήθησε πάρα πολύ να εξελιχθούν οι διάφορες ε, πολιτιστικές πολιτικές. Ε, μιλάμε για το μέλλον της πολιτιστικής πολιτικής. Όταν ξεκίνησε η διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέλλον της Ευρώπης, ε, θελήσαμε να δούμε ότι συμπεριλαμβάνεται και ο πολιτισμός. Και ένα χρόνο μετά βλέπουμε ότι όντως Τι κάναμε λοιπόν. Ξεκινήσαμε διαβουλεύσεις. Από τις μεγαλύτερες διαβουλεύσεις για το τι μπορεί να προσφέρει ο πολιτισμός στο μέλλον της Ευρώπης και πώς πρέπει να εξελιχθούν οι μελλοντικέ πολιτικές της Ευρώπης για τον πολιτισμό. Δημιουργήσαμε λοιπόν 8 ευρωπαϊκούς κόμβους, σε 8 δηλαδή διαφορετικές χώρες, όπου συμμετείχαν 527 άνθρωποι, οι οποίοι συμμετείχαν σε μια συζήτηση σε μια συνομιλία για το μέλλον ε, του πολιτισμού στην Ευρώπη και καταλήξαμε σε έξι κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες μπήκαν σε μια ψηφιακή πλατφόρμα. Αυτές οι έξι κατευθυντήριες γραμμές ποιες είναι λοιπόν αποτελούν και το περιεχόμενο του εγγράφου μας για το μέλλον του πολιτισμού και μπορεί κανείς ε, να τη συμβουλευτεί. Μπορούμε λοιπόν, πιστεύουμε, μετά τις διαβουλεύσεις να παρουσιάσουμε μια σαφή εικόνα του τι θέλει ο κόσμος και ποιες είναι οι έξι κατευθυντήριες γραμμές. Πρώτον, χρειαζόμαστε μια ισορροπημένη και ανοιχτή προσέγγιση απέναντι στον πολιτισμό. Προηγουμένω όμως θα έλεγα ότι δεν έχουμε σημεία αναφορά όσον αφορά την ε, δημιουργία και την πολιτιστική κληρονομιά που αποτελούν και την βάση. Θα έπρεπε να είναι να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Λοιπόν, ισορροπημένη προσέγγιση είπα. Είναι βέβαια δύσκολο, πράγματι. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει επιθυμία για κάτι τέτοιο, για να πετύχουμε αυτή την ισορροπία. Βέβαια, οικονομικός πυλώνας είναι αυτός ο οποίος υπερισχύει. Παρόλο που υπάρχουν και ανοίγματα, να υπάρχουν ε, δίκες αμοιβέ, για παράδειγμα, μέσα σε αυτό το οικοσύστημα. Βλέπουμε να συμπεριλαμβάνεται η εκπαίδευση. Πρέπει να δούμε ο πολιτισμός και η εκπαίδευση τι ρόλο παίζουν. Η εκπαίδευση βέβαια είναι κάτι γενικότερο οικονομικά. Όμως εμείς βλέπουμε εγκάρσια προσέγγιση. Πολιτιστική κληρονομιά. Όπως έχουμε ξαναπεί, είναι σημαντικό, όπως μας έδειξε η διάσκεψη για την πολιτιστική κληρονομιά, ότι υπάρχει και η ζωντανή κληρονομιά. Πρέπει να υπάρχει σύνθεση ανάμεσα στην ε, πολιτισμική κληρονομιά και την σύγχρονη δημιουργία. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία δηλαδή ανάμεσα στις ε, υποδομές παντοσίδους. Τώρα για την τομιακή προσέγγιση. Εδώ θα επαναλάβω αυτό που είπε και ο κ. Βακέλα, ότι δηλαδή στις διαβουλεύσεις βλέπουμε ότι στις ε, δράσεις, την όλο και μεγαλύτερη βρυδιακή μορφή του πολιτισμού. Βλέπουμε ότι οι συνέργειες αποκτούν και όλο μεγαλύτερη σημασία, όμως βλέπουμε ότι έχει διαφορετική προσέγγιση η ατζέντα. Άνηση αντιμετώπιση βέβαια οδηγεί και στην πολυμορφία που σας έδειξα πριν με τις περίεργες διασυνδέσεις. Όμως ένα από τα βασικά στοιχεία είναι η πολιτιστική διάσταση των σημερινών εξελίξεων κοινωνικών και άλλων εξαιτία τη μετανάστευση που απασχολεί τόσο πολύ την Ευρώπη. Συζητήσαμε λιγάκι ότι υπάρχει διχοτομία. Ε, την μια μεριά η πολυμορφία, πολιτιστική, από την άλλη μεριά ο διάλογος και δυνατότητα συμμετοχής όλων στον πολιτισμό. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις πρέπει να συνδυαστούν. Ξέρουμε ότι όσοι ασχολούνται με τον πολιτισμό συμμετέχουν περισσότερο σε πολιτιστικές ε, πρωτοβουλίες, τους ενδιαφέρει ευημερία κλπ. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια συνολική προσέγγιση. Για την κινητικότητα τώρα. Πολλά έχουν υποθεί μέχρι τώρα. Η πρωτοβουλία αυτή είναι ευπρόσδεκτη βέβαια. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμεί θα θέλαμε να είναι πραγματικά φιλόδοξη και για το πεδίο εφαρμογή, ώστε να συμπεριληφθούν παντό είδου δημιουργοί, οι ίδιοι δημιουργοί, οι οργανώσει του κλπ. Αλλά και στην οικονομική στήριξη να είναι επίση φιλόδοξη η Επιτροπή. Τώρα, όταν είχαμε τι διαβουλεύσει αυτές, μια από τις εγκάρσιες εξελίξεις είναι ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες δυσκολίες για την ελευθερία έκφρασης των δημιουργών στην Ευρώπη. Για χρόνια δεν αντιμετωπίσαμε αυτό το ζήτημα καθόλου. Ξεχάσαμε πώς να δράσουμε γι' αυτό. Και τώρα δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι θα έπρεπε να στηρίξουμε τους δημιουργούς, τις οργανώσεις τους, να ξέρουν ποια είναι τα δικαιώματά τους, να ξέρουν πώς μπορούν να αντιδράσουν άπαξ και γίνουν θύματα επιθέσεων. Και αυτό σε συνεργασία με τον Οργανισμό για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία να είναι ευαίσθητα σε αυτό το ζήτημα. κυρίως στα πλαίσια της σύγχρονης ε, έρευνας για τη δημιουργία. Βλέπουμε ευτυχώς ότι συμπεριλαμβάνεται η εκπαίδευση στους στόχους του πολιτισμού. Και είναι καλό. Πρέπει επίσης να υπάρχει συνέργεια ανάμεσα στην εκπαίδευση και την ε, δημιουργία αλλά και την καλλιτεχνική έρευνα. Θέλουμε ενίσχυση του διαλόγου. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε μόνο και να τονίζουμε μόνο την ευρωπαϊκή διάσταση του πολιτισμού. Έπειτα πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι οι τομείς πολιτισμού και έρχομαι και στο τελευταίο που είναι η συλλογή δεδομένων. Υπάρχουν οι ψηφιακές πλατφόρμες που έχουν τα πάντα. Από την άλλη έχουμε το δημόσιο τομέα, ο οποίος δεν έχει τόσα πολλά δεδομένα. Χρειάζεται λοιπόν συνεργασία και να ξέρουμε ότι η συλλογή δεδομένων δεν θέτει σε κίνδυνο τα οικονομικά δεδομένα. Και αυτό είναι κάτι ζωτικής σημασίας για το μέλλον. Μίλησα πριν για φιλόδοξους στόχους. Όντως, χρειαζόμαστε φιλοδοξία και στην οικονομική στήριξη. Η Culture Action Europe ζητάει διπλασιασμό των κονδυλίων για την Ευρώπη και εκατό στο κάθε πολιτιστικό κλάδο. Ευχαριστώ πολύ. Ja, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεισφορά σας στην συζήτησή μας. Κοιτάω ποιος θέλει. Σίλβια Κώστα, δύο λεπτά. Συνοπτικότατα, να πω ότι εκτιμώ πολύ τη δουλειά σας εδώ και πολλά χρόνια. Έχετε οργανώσει επανειλημμένους ε, διαβουλεύσεις. Έχω δει αυτές οργανώσετε και στη χώρα μου και ήταν πολύ καλές. Είναι τρία τα σημαντικά στοιχεία στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε. Πρώτον, ότι χρειάζεται περισσότερη παρουσία και ε, υπογράμμιση τη δημιουργική ε, διάσταση, όπω υπόθηκε προηγουμένω. Αυτή πρέπει να προωθηθεί. Συμφωνώ με το ε, δεξιότητε για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Πρέπει να γίνει σωστή διασύνδεση και την οπτική γωνία, όχι μόνο των STEM αλλά και των STEAM. Και Κάτι που είπε προηγουμένω και ο Ούγκο Μπακέλα. Αυτά που προσδοκούμε ως κληροδότημα και από το Ευρωπαίο και ο που ήταν ε, ορόσημο για πολλά πράγματα. Και το να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση, αλλά και διατομιακή διεπιστημονική. Μια διακυβέρνηση με μεγαλύτερη συμμετοχή. Μια διαχείριση με μεγαλύτερη συμμετοχή. Αυτό και για το πρόγραμμα διά, ε, δράσης που θα ακολουθήσει, σημαντικό είναι να μην χάσουμε αυτή τη διαχείριση, την governance, που ήταν μια από τις επιτυχίες του ευρωπαϊκού έτους, με τις διαβουλεύσεις σε τόσα πολλά επίπεδα και με τόσους πολλούς ε, stakeholders, συμμετέχοντες να ε, είναι στο παιχνίδι. Ευχαριστώ. Θέλετε να απαντήσετε αμέσω, παρακαλώ. Yes, uh... Ναι. Συμφωνώ πόσο μεγάλη σημασία έχει ο πολιτισμός να λαμβάνεται υπόψη σε όλες ε, τις πολιτικές. Όταν κοιτάμε άλλα προγράμματα βλέπουμε ότι επιλέγονται κάποιοι τομείς ή μόνο κερδοσκοπικός ε, χαρακτήρας. Οπότε αν θέλουμε να είμαστε επιτυχείς στον επόμενο κύκλο των προγραμμάτων πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ολόκληρο τον ε, κλάδο της πολιτιστικής δημιουργίας και να υπάρχει mainstreaming. Δηλαδή να λαμβάνεται υπόψη ο πολιτισμό σε όλε τι πολιτικέ. Είναι πολύ βασικό για το μέλλον, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χέλγα Τρίπελ. Ναι, εγώ θα ήθελα να έρθω στο θέμα της συλλογή των δεδομένων και της ανισορροπίας μεταξύ ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα των αμερικανικών τεχνολογικών ε, γιγαντών και την έλλειψη που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Ξεκίνησα μόνιμο ζητώντας τον επόμενο προϋπολογισμό να ζητήσω μια ευρωπαϊκή δημόσια ψηφιακή πλατφόρμα. Και δεν ξέρω, πριν από 10 χρόνια δεν τα καταφέραμε και τώρα ξαναξεκινήσαμε τη συζήτηση να μην τα αφήσουμε στα ιδιωτικά μονοπόλια, κάτι το οποίο βεβαίως είναι δύσκολο να ελέγξουμε και να επηρεάσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω εάν το συζητάτε εσείς αυτό το θέμα περί μιας πανευρωπαϊκής πλατφόρμας με προστασία δεδομένων, με άδεια χρήσης του περιεχομένου και πρόσβαση για τον Ευρωπαίο πολίτη. Τι άποψη έχετε γι' αυτό. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Πέρες, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Πολύ επίκαιρη. Εμείς ε, στην Τίμη Σοάρα, στην διάσκεψή μας τον Οκτώβριο ακριβώς ασχοληθούμε με τα ψηφιακά ζητήματα ε, και είστε φρόσδεκτοι βεβαίω. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν ψηφιακές ε, πολιτιστικές κοινότητες αλλά δεν είναι συνδεδεμένες. Δεν έχουμε λοιπόν την κλίμακα τον όγκο και αυτό είναι ακριβώς ένα ερώτημα που θα συζητηθεί στην διάσκεψη αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Σόντροβα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε που δεν ήμουν εδώ από την αρχή. Έπρεπε να είμαι και στην Επιτροπή Επασχόληση δίπλα. Αλλά ευχαριστώ για τι ε, παρουσιάσει σα και τι ομιλίε σα. Άκουσα στην τελευταία παρουσίαση κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα για την ευρωπαϊκή πολιτική πολιτισμού. Λόγω χάρη, μπορείτε να μας πείτε τη γνώμη σας ή να μας δώσετε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμβαίνουν πολλά πράγματα θαυμάσια, υπέροχα, όπως τα βραβεία ή οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες. Ε, μια δεκαριά πόλεις ήδη έχουν αξιοποιηθεί διαφορετικά. Ε, το πρώτο. Το δεύτερο, τα μνημεία. Τα μνημεία τα οποία έχουν μπει στο ε, heritage. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά με εκθέσεις, αναπαράσταση και ούτω καθεξής. Τα μνημεία αυτά η παρουσίαση τους θα είναι καλό να συνεχιστεί ε, να υπάρξει κάποιο είδους ε, διαδικτύωση, κάποιο είδους συνέχεια με κοινή δουλειά. Αλλά χρειάζεται και ευρωπαϊκή στήριξη με το Creative Europe ας πούμε. διότι τώρα δεν στηρίζονται. Δυστυχώς λοιπόν νομίζω ότι ε, δεν είμαστε αρκετά αποτελεσματικοί σε σχέση με το χρόνο και την ενέργεια που χρειάζεται. Πρέπει να αξιοποιήσουμε ότι έχει ήδη γίνει πρώτα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να υποστηρίξουμε τα πραγματικά παραδείγματα καλής εργασίες ε, για τον πολιτισμό σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και εθνικό. Ευχαριστούμε κυρία Πέρες. Ευχαριστώ. Υπάρχουν δύο διαστάσεις στην ερώτησή σας. Ειλικρινά, στον πολιτιστικό τομέα δεν βρίσκουμε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο το θέμα αυτό το βραβείο. Τώρα η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα είναι το αντίθετο. Είναι μια μεγάλη στήριξη όλων των πρωτοβουλειών. Και γίνεται πολλή δουλειά σε τοπικό επίπεδο. Η δεύτερη διάσταση έχει να κάνει με τη διακυβέρνηση, την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Αυτό είναι κάτι που αποκτάει όλο και μεγαλύτερη σημασία. Ίσως δεν κάνουμε αρκετά για να τα συνδέσουμε όλα αυτά τα επίπεδα. Θα πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση γιατί είναι ο μόνος τρόπος να υποφεληθούμε όσο γίνεται περισσότερο από τον ευρωπαϊκό πολιτιστικό χώρο. Για μια συγκεκριμένη πτυχή διακυβέρνησης που έχει να κάνει με την πολιτιστική κληρονομιά, από τις πιο επιτυχείς διαστάσεις είναι ακριβώς η ομάδα των εταίρων. Γιατί βλέπουμε ότι εκεί υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, πολύ κλάδη και η πρότασή μας είναι να διατηρηθεί και πέρα το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για να σκεφτούμε μαζί πώς μπορεί να υπάρξει συνέχεια με το ίδιο πνεύμα που μας φέρνει πάλι στην ιδέα της διακυβέρνησης που πρέπει να είναι σε συνεργασία με τους χώρες μέλη, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με μια προσέγγιση δηλαδή ανοιχτή υπέρ της συμμετοχής όλων. Παρακαλώ. Ε, και σύντομα, αν γίνεται. Θέλω να προσθέσω κι εγώ κάτι, παρακαλώ, στο θέμα της διακυβέρνησης και εταιρική σχέσης συνεργασίας. Αν πραγματικά θέλουμε να φέρουμε τον πολιτισμό σε κεντρικό σημείο και να μην είναι στο περιθώριο, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλους τους παράγοντες του πολιτιστικού οικοσυστήματος. Δηλαδή, όχι μόνο τη διανομή και την παραγωγή πολιτισμού, αλλά και τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών, τα θεμέλια και τις τοπικές αρχές, παντού. Και νομίζω ότι Κάτι εδώ θα μπορούσε να αναπτυχθεί παρετέρω. Η πρόθεση, η στήριξη των τοπικών περιφερειακών εταίρων. Μαζί τους να δουλέψουμε, να δούμε τι πετυχαίνει και τι πετυχαίνει λιγότερο σε τοπικό επίπεδο. Αυτό θα μπορούσε να συνεισφέρει πάρα πολύ καλά ε, στην Ευρώπη υπέρ ευρύτερων συμμαχιών. Αυτή είναι η εγγύηση, πιστεύω, για το μέλλον του πολιτισμού, πέρα από τις δημόσιες πολιτικές βέβαια. Επίσης, ας σκεφτούμε και την σχέση ε, και την, ε, τα όσα κάνουν ε, τα ιδρύματα. Υπάρχουν πολλά ιδρύματα και στην Ιταλία και την Πορτογαλία και τη Γερμανία και αλλού πάρα πολλά ιδρύματα τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα. Καινοτόμα πραγματικά. Το τάντεμ και πολλά άλλα. Ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και μικρά πιλωτικά προγράμματα. Θα πρέπει να δούμε σε αυτά τα προγράμματα τι λειτουργήσε καλά και να το λάβουμε υπόψη μας σε άλλα προγράμματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το οποίο μας είπατε και για τα ιδρύματα. Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε και το ίδρυμα στην ε, Λισαβόνα και είδαμε πολλά από τα ε, έργα ευρωπαϊκού τύπου και καλλιτεχνικών ανταλλαγών και νομίζω ότι ε, είναι πάρα πολύ το, κάτι το πάρα πολύ θετικό. Η κυρία Τζούλι Γουόρτ. Πρώτα απ' όλα να πω ότι χαίρομαι που βλέπω την Ρόζα. Εγώ είμαι μέλος της Culture Action Europe. Μπορείτε να γίνετε μέλη και θα σας έλεγα να γίνετε. Εγώ πηγαίνω ε, εκεί στις διασκέψεις, όχι ως πολιτικός, αλλά ως ε, μέλος. Ε, ήμουν και από πριν μέλος και θα είμαι μετά. Και είναι νομίζω κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε. Και Βεβαίω ε, θεωρώ ότι τέτοιες οργανώσεις θα ε, πάνε καλά γιατί αντιλαμβάνονται την ολιστική φύση του πολιτισμού ε, ότι εμπλέκεται σε διάφορους τομείς της ζωής. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό, αλλά η δυσκολία είναι όταν σκεφτόμαστε έτσι μεμονωμένα ο καθένας και στο επίπεδο της ε, Κομισιόν. Τα είχαμε πάει λοιπόν πολύ καλά με την πολιτιστική διπλωματία και με την Επιτροπή των Εξωτερικών. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω τι θεωρείτε ότι πρέπει να κάνουμε κατόπιν για να προωθηθεί αυτή η πολιτική. και Βεβαίω, βλέπουμε τις διαφορές προσπάθειες να συνδυάσουμε τις τέχνες με τις θετικές επιστήμες, όχι μόνο θετικές επιστήμες. Αν μιλήσουμε λοιπόν για προτεραιότητες ε, που πρέπει να δώσουμε την μάχη για να αναγνωριστεί ο, ο πολιτισμός από τους άλλους κλάδους. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως που είστε μέλος μας. Ναι, πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Πρέπει ακριβώς ε, να προχωρήσουμε, προχωράμε δηλαδή, αλλά δεν υπάρχει ακόμα μια συνεκτική πολιτική, κάπου ακουστήμ, κάπου ακουστέμ. Δηλαδή κάπου έχουμε τις θετικές επιστήμες, κάπου είναι οι τέχνες εντό παρενθέσεως και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Ε, τώρα όσον αφορά τους άλλους τομείς πολιτικής, εγώ θα έλεγα ότι ένα θέμα είναι η πολιτική συνοχή. Έχουμε το πρόγραμμα ΕΤΠΑ όπου κοιτάμε την συμπερίληψη του πολιτισμού γιατί βεβαίως θεωρούμε ότι θα έπρεπε να περιληφθεί ένα στόχος ειδικά για τον ε, πολιτισμό και η άλλη διάσταση είναι η έρευνα, η έρευνα και η καινοτομία και το πρόγραμμα ε, ορίζοντας ε, όπου έχει αρχίσει να αναγνωρίζει τον πολιτισμό αλλά η καλλιτεχνική έρευνα πρέπει να την δούμε στο ίδιο επίπεδο με την επιστημονική έρευνα. Βλέπουμε εντάξει την ψηφιακή οικονομία που την ανέπτυξαν μηχανική. Εμείς ξέρουμε όμως ότι της λείπει μια κοινωνική διάσταση για να λειτουργεί. Πρέπει λοιπόν να το αναγνωρίσουν αυτό επίσης όρις. Εγώ εκεί θα επικεντρωνόμουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ να ακούσουμε και τον κύριο Σαμπιέρη από την Κομισιόν για τρία λεπτά παρακαλώ. Thank you very much. Um, and Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή που δίνετε στο εγγραφό μας. Ε, εντάξει, δεν θα έλεγα ότι εκπλήσωμαι, αλλά πάση περιπτώσει ο βαθμός λεπτομέρειας με τον οποίο ενημερωθήκατε, ναι. Η στόχη αυτή ξεκινούν από το γεγονός ότι οι πολίτες εμπιστεύονται τη δύναμη του πολιτισμού γενικά στην Ευρώπη. Αλλά συγχρόνως διαπιστώνουμε ότι για πολλούς ε, Ευρωπαίους οι χώρες μέλη διαφέρουν όσον αφορά τις αρχές και τις αξίες. Και πολύ σωστά είπατε ότι πρόκειται για τους στόχους που αναφέρονται στις ε, ικανότητες των ατόμων. Δηλαδή δεν πρόκειται για την καινοτομία, πρόκειται για τους καινοτόμους πιο πολύ. Τι μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν. Και αυτό εξηγεί και κάποιες επιλογές που έχουμε υιοθετήσει. Το γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η κινητικότητα θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της οικονομία βεβαίως, γιατί υπάρχουν οικονομικές συνέπειες από την κινητικότητα εννοείται. Και θα μπορούσαν να υπάρχουν και κοινωνικοί στόχοι. Αλλά αν διαβάσετε προσεκτικά θα δείτε ότι εμείς ό,τι προτείνουμε για την οικονομική διάσταση είναι η δημιουργία μέσα στην οικονομία. Γιατί θέλουμε να είμαστε μια ήπειρος δημιουργίας. Γιατί πιστεύουμε ότι η δημιουργία μπορεί να έχει πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Στη χημεία, στις επιστήμες γενικά. Και γι' αυτό θέλουμε και έναν ευρύτερο ορισμό της οικονομίας και όχι μόνο ότι είναι ο αριθμός ε, της απασχόλησης ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τον πλούτο των καλών ειδών. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτιστική κληρονομιά και το θέμα της συμμετοχής είναι τα βασικά ζητήματα στις προτάσεις μας. Και υπήρχαν και στην ανακοίνωσή μας του 2014 τότε για το Ευρωπαϊκό Έτος. συνεχίζουμε να τα βάζουμε στο κέντρο του προβληματισμού μας και των προσπαθειών μας. Η συνοχή τώρα ανάμεσα στις εσωτερικές και τις εξωτερικές πολιτικές έχει πολύ σημασία και για μας. Το τονίζουμε στην κοινή μας ανακοίνωση πριν από δύο χρόνια και ακριβώς την ίδια μεθοδολογία προτείνουμε τώρα στη σχέση μας με τις χώρες εταίρους αλλά και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες μέλη είναι ο πολιτισμό αρμοδιότητα των χωρών μελών στο κάτω-κάτω, αλλά οι στόχοι αυτοί αποτελούν την πρότασή μα και προς τις χώρες μέλη, προκειμένου να συνεργαστούμε για κάποια συγκεκριμένα προγράμματα. Και αυτό προτείνουμε ε, πώς συμμετέχει ας πούμε ο πολιτισμός στην κοινωνία, η καινοτομία. Εγκρίνοντας τη μεθοδολογία αυτή ήταν πιο εύκολο για μας να βρούμε και χώρο για τον πολιτισμό στα διάφορα προγράμματα που προτείνουμε. Είναι πιο εύκολο να συζητούμε με τα Υπουργεία αν μπορούμε να το πούμε εμείς τι μπορούμε να προσφέρουμε. Και όπως γίνεται πάντα και εδώ πρέπει να σας πω ότι το θέμα της ε, ποιότητας της τέχνης βέβαια δεν ε, έχει την ίδια θέση. Εντάξει, μπορεί να είναι κάποια παραβίαση της επικουρικότητας. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξή σας στις επιλογές μας, όπως για παράδειγμα στην κινητικότητα. Σας είμαστε ευγνώμονες και ελπίζουμε να συνεχιστεί ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν βεβαίω όπω φέρει κανεί λεφτά, αυτομάτω βελτιώνεται η ατμόσφαιρα. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Θα ήθελα να, δώσω τον, να ρωτήσω τον κύριο Γραμματικά και αν θέλει να πει κάτι για δύο λεπτά. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και οι τρεις συγγύσει ε, και πραγματικά, κυρία Πρόεδρε, θέλω να επενέσω τους συγγητές γιατί έδωσαν πολλές φορές και νέες διαστάσεις ε, στο μεγάλο αυτό θέμα της του ευρωπαϊκού πολιτισμού και με εντυπωσίασαν ιδιαίτερα. Θα κάνω μόνο μία παρατήρηση. Νομίζω αυτό που αναφέρθηκε από πολλούς ομιλητές ότι δεν πρέπει να επιδιώκουμε κατά κάποιο τρόπο ένα χρήσιμο, χρησιμοποιώ μια λέξη πρόχειρα, το, μόνο το χρήσιμο πράγμα στον πολιτισμό, δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό χαρακτηρίζει και τη σημερινή ευρωπαϊκή παιδεία. Ε, και νομίζω αυτή είναι η αιτία του κακού. Δηλαδή η ευρωπαϊκή παιδεία, η παγκόσμια παιδεία, αυτή τη στιγμή αποφεύγει να δημιουργήσει ανθρώπους ολοκληρωμένους, περίεργους, ανήσυχους, ανικανοποίητους και κυρίως κατευθύνει τα νέα παιδιά, το ξέρω από τη δική μου εμπειρία, στο τι είναι χρήσιμο στην επιστήμη ή ακόμα περισσότερο το τι έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να κερδίσει πολλά χρήματα. Αυτό νομίζω επηρεάζει πάρα πολύ, η παιδεία επηρεάζει πάρα πολύ και την γέννη κατάσταση του πολιτισμού και εκεί βλέπεις παρόμοια φαινόμενα και ελπίζω να βρούμε τρόπους να το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ και πάλι πολύ όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσατε τους επένους. Νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι. Χαίρομαι που ήσασταν σήμερα εδώ. Νομίζω ότι ήταν σημαντική η συνεισφορά σας ε, για την περαιτέρω εργασία και για την ατζέντα του πολιτισμού αλλά και ε, βεβαίω όλα αυτά σχετίζονται τελικά με το πρόγραμμα Creative Europe το οποίο μας απασχολεί αυτή την στιγμή, με αυτό εργαζόμαστε. Και ελπίζω να υπάρξουν οι βελτιώσεις ε, σε αυτά τα οποία προτείνονται. Μας δώσατε λοιπόν πολλά ερεθίσματα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και ε, καλή επιστροφή εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα ε, έχω να σας ανακοινώσω ότι η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 3 Σεπτεμβρίου από τις 3 μέχρι τις 6.30. Επιπλέον. Σας εύχομαι ωραιότατο καλοκαίρι. Νομίζω πραγματικά το κερδίσαμε, το αξίζουμε, εργαστήκαμε πολύ τους τελευταίους έξι μήνες ε, και το επόμενο εξάμεινο και μέχρι τις ευρωεκλογέ ε, θα είναι επίσης εντατικό, οπότε ξεκουραστείτε, βρείτε τους οικείους σας και θα τα ξαναπούμε στις 3 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε καλά να είστε. Το ίδιο ισχύει και για τους ε, διερμηνείς. Ε. Ευχαριστούμε και εμείς την Πρόεδρο. Και καλό καλοκαίρι σε όλους. Ευχαριστώ. Θα ε, γίνει αμέσως μετά η συνεδρία των συντονιστών.